Ε, τι θέση, τι πιστεύετε, ποια γνώμη έχετε, ώστε να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Έχουμε ακόμα δυόμιση χρόνια στα οποία δεν θα μας απασχολήσει σχεδόν τίποτα άλλο παρά αυτές οι εκθέσεις. Άρα μία κατά την ε, πάυση των Χριστουγέννων να σκεφτούμε την κατανομή των εκθέσεων αυτών. Και θα αποφασίσουμε, θα αποφασίσουμε στην αρχή τη συνεδρίαση των συντονιστών για να μην ξανασυναντηθούμε το Δεκέμβριο και να αλλάξουμε πάλι όλα τα πράγματα και να πούμε όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο. αύριο το πρωί ε, ένας συνάδελφός μας θα μιλήσει για τις απονομές ε, του βραβείου Λουξ. Αλλά αυτά αύριο το πρωί. Τώρα, σημείο 4, σήμερα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς. Ε, πιστεύω ότι αυτό υπό την Ουγγρική Προεδρία το έχουμε συζητήσει ενδελεχώς. Η κυρία Παλιαδέλη τα διαχειρίστηκε όλα θαυμάσια. Όμως οι διαδικασίες αργούν, αργούν και δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Το Συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει, τώρα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο και έτσι στην επόμενη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μπορούμε να το διευθετήσουμε χωρίς καμία, κανένα πρόσκομα. Η κυρία Παλιαδέλη έκανε μια εξαιρετική διαπραγμάτευση εξ ονοματός μας και είχαμε <laughs> μία θαυμάσια συνεδρίαση όπου και οι δύο τσακωθήκαμε πάρα πολύ καλά. Η κυρία Παλιαδέλη έχει το λόγο. Yes, you do. So I'll read my English text. Θα σας διαβάσω το κείμενό μου στα αγγλικά Πέρα από την αρχική μου πρόταση για την αλλαγή του τίτλου για το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομίας, για το οποίο δεν κατάφερα να πείσω βέβαια τους σκιώδους ηγητές, ουσιαστικά μέσω των τροπολογιών προσπάθησα να διασαφηνίσω κάποια ζητήματα τα οποία ήταν ασαφή στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που τελούν εγγύηση για την διατήρηση του νέου αυτού θεσμού του σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιά Πρώτον, ο αριθμό των χώρων που θα μπορούν να πάρουν το σήμα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Δεύτερον, και έπειτα η συνέχεια ανάμεσα στην διακυβερνητική πρόταση και την επίσημη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήξαμε έτσι σε ένα τελικό κείμενο το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή μα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια στη συνέχεια και αποτελεί πλέον σημείο αναφορά για τη συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια πρώτη φάση το σήμα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά ήταν ανοιχτό για τη συμμετοχή των κρατών μελών μόνο, όχι μόνο όπως ε, είχε, όχι όπως είχε υποθεί στην αρχή, δηλαδή για τη συμπερίληψη και τρίτων κρατών μελών. Στη συνέχεια βέβαια θα εξεταστεί αν πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογή. Δεύτερον, η επιλογή των χώρων θα γίνεται κάθε δύο χρόνια και όχι σε αιτήσια βάση, προκειμένου να αποτρέψουμε να έχουμε μια πολύ έντονη αύξηση του αριθμού των χώρων που μπορούν να πάρουν το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς. Τρίτον, όταν έχουμε πολλούς χώρους επιλέξιμου στα πλαίσια ενός, ενός κράτους μέλους, τότε στην περίπτωση αυτή καλούνται οι χώροι αυτοί να συνεργαστούν μεταξύ τους και να υποβάλουν μία ενιαία αίτηση. Αυτό είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου, με συγχωρείτε, το οποίο ενέκρινε και η δική μας Επιτροπή. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Στο αρχικό κείμενο χρησιμοποιήσαμε τον όρο διακρατική χώρη και αυτό έχει αποσαφινιστεί. Το ζήτημα των ποσοστώσεων ουσιαστικά επιλύεται σε επίπεδο κράτους μέλους τώρα. Επιλέχθηκε η λύση αυτή για να μην έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης, αλλά και για να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στις συνδυασμένες αυτές αιτήσει, οι οποίες συμβάλλουν στο να ενδυναμωθεί η κοινοτική συνοχή. Τέλος, οι μεταβατικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με τους χώρους που έχουν ήδη εγκριθεί από τη διακυβερνητική πρωτοβουλία στο αρχικό κείμενο οι σχετικές διατάξεις ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκες και ουσιαστικά επέβαλαν διαφορετικά κριτήρια από αυτά τα οποία προβλέπονται στη νέα δράση. Η δική μας πρόταση για να διαγραφούν τα αρχικά κριτήρια οδήγησε τελικά σε έναν επικοδομητικό συμβασμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τελικά καταλήξαμε σε ένα πολύ πιο σύντομο και απλοποιημένο σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα τα σχετικά, θα εξεταστούν τα αρχικά κριτήρια της ε, διακυβερνητικής πρωτοβουλίας, όσον αφορά την επιλογή των νέων χώρων και θα ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή και για τις νέες αιτήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού που μου ανέθεσαν αυτή την τόσο σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω όμως και τους κοιόδης ηγητής για την επικοδομητική του συνεργασία, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Να ευχαριστήσω επίσης το διοικητικό προσωπικό και το νομικό προσωπικό για την επιτυχία της όλης διαδικασίας, την Βελγική Ουγγρική και Πολυλονική Προεδρία για, την ιδιαίτερη, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο δείξανε προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Και τέλος την ε, πρόεδρό μα, την κυρία Ντόρι Πακ, για την παρουσία της και τη συμβολή της στο τελικό αυτό θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. So, is there any... Anybody of the... Υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Yes, Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κυρία Παλιαδέλη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει σε ένα πολύ θετικό συμβασμό με το Συμβούλιο και προσβλέπουμε πλέον στην επίσημη έγκριση του κειμένου το συντομότερο δυνατό και ελπίζουμε να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα η σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Πιστεύω πραγματικά ότι ε, θα έχει την ίδια αξία στο μέλλον όσο και οι πολιτιστικές ε, πρωτεύουσε. Κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και στις ε, αρχές του επόμενου έτου, θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία προκειμένου να επιλεγούν οι χώροι αυτοί για το 2013. Ευχαριστούμε και οδησηγήτρια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω την κυρία Παλιαδέλη γιατί πραγματικά έδειξε πάρα πολύ μεγάλο σθένος προασπιζόμενοι τα σημεία αυτά τα οποία θέλαμε να διατηρήσουμε. Τα σημαντικά αυτά σημεία έχουν να κάνουν με την απλοποίηση καταρχάς της όλης διαδικασίας προκειμένου να καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να πετύχουμε και έπειτα όσον αφορά τα σαφή αυτά κριτήρια τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε, τα οποία πρέπει να συνάθουν με τους βασικούς μας στόχους και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το κατάλληλο σύστημα επικοινωνία, προκειμένου τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να καταλάβουν την όλη διαδικασία και να μπορούν να συμβάλλουν στην προάσπιση τη ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια. προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε ένα επιτυχημένο σύστημα στα πλαίσια του σήματο Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Είχαμε μια πολύ καλή επικοδομητική συνεργασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συμφωνούμε στι βασικέ αξίε του ζητήματο αυτού. Τζον Κέλλη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τους προλαλήσαντες. Απλώς είμαι λίγο απογοητευμένος ε, που δεν άλλαξε ο τίτλος. Ε, γιατί πιστεύω ότι ε, το σήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική προνομίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και, και άπτεται ακριβώς του μεγάλου θέματος του ευρωσκεπτικισμού των αρνητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ε, ο στόχος είναι προφανής να δημιουργήσει και να προβάλλει την Ευρωπαϊκή Ενότητα και ε, έχει μια συμβολική αξία ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι η ιδέα της, του, του, μιας ε, διετούς ε, αξιολόγησης είναι πάρα πολύ καλή και όχι ετήσιας. Δηλαδή αυτό το διετές πλαίσιο είναι σωστό. Και επίσης η, επιλογή ενός εθνικού θέματος, μια εθνικής ε, θεματικής ενότητας, η επιλογή πολλαπλών χώρων είναι επίσης πολύ σωστή ιδέα. Είμαι απογοητευμένος που η δική μου η χώρα δεν το έχει ακόμα υποστηρίξει, δεν το έχει υιοθετήσει, αλλά πιστεύω ότι ακολουθούμε ένα πολύ σωστό δρόμο. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι που υποστηρίζουν αυτό το θέμα και που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά θέματα ε, θα ασκήσουν πίεση για να ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το δρόμο για να το επικυρώσουμε. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι πιστεύω να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την απόφαση. Ε, η Πρόεδρος, Ευχαριστώ. Παρόλο που δεν λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, το σήμα θα έχει ε, το, το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ανησυχείς, θα υπάρχει οπωσδήποτε αναφορά και θα, θα δείχνεται και στο σήμα. Ε, άλλος κανείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτές τις πολύ σημαντικές συστάσεις. Νομίζω ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στις περισσότερες επιφυλάξεις και ανησυχίες μας με αυτό το λίγαν εμπεριστατωμένο και πολύ ενδιαφέρον κείμενο που έχουμε. αναφέρεται σε, όλες αυτές τις θεματικές ενότητες, τις διακρατικές ε, τοποθεσίες. Ε, ε, επίσης αυτό το δείχνει μία πορεία που ξεπερνάει εθνικά σύνορα. Αυτό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας, της ενότητας της Ευρωπαϊκής Υπήρου και πιστεύω ότι αυτό, αυτή η θεματική ενότητα πρέπει να καλύπτει και το θέμα της διάστασης του φύλου. Πρέπει να υπάρχει μια ισότητα στην ε, μεταχείριση των φύλων και σε αυτό το θέμα. Και επίσης να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα η αρχή της επικουρικότητας. Ιδίω ε, στην επισήμανση των τοποθεσιών από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δεσμεύσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουν η αναζήτηση καταλήλων και επιλέξιμων τοποθεσιών ε, θα, θα εμπλέξει και τα πανεπιστήμια, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώσεις πολιτών και γενικά όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να γνωρίζω πόσα κράτη βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα αυτό για το σήμα. Μπορεί κάποιος να μου πει πόσα κράτη είναι ήδη στο σύστημα αυτό. Ναι. Αυτό είναι μία, ένα καινούριο σήμα, έτσι. Αλλά ε, είναι μία συνέχεια του ήδη υπάρχοντος. Άρα ορισμένα κράτη-μέλη ήδη συμμετέχουν, πολλά όμως όχι, διότι δεν είναι μία αυστηρά δομημένη υπόθεση αυτή. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας φωτίσει για τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν μπορώ. Ε, μικρόφωνο παρακαλώ. Εάν θυμάμαι καλά, κατά την διακυβερνητική ήταν 64. Τώρα θα εφαρμοστεί κατά την πρώτη εφταετή περίοδο στα κράτη-μέλη μόνο. Εν συνεχεία θα κάνουμε μία αναθεώρηση για τη συμμετοχή ή όχι τρίτων χωρών σε αυτό το σήμα. Θα δεχτούμε δηλαδή υποβολή αιτήσεων για το σήμα. Κομισιόν, πόσες χώρες παρακαλώ, ξέρετε. Ναι, όπως είπατε, ε, βάση, ε, υπό τη διακυβερνητική ήταν 64 χώροι, 64 χώροι και 17 χώρες. Αλλά με το νέο σχέδιο θα πρέπει να γίνει επανεξιολόγηση με τα νέα κριτήρια. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα παρακαλώ σε αυτό το θέμα. Αν όχι τότε προχωρούμε στο 5. ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Και ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα αυτό βεβαίως βασίζεται στις καινοτομίες, στην πολυπολιτισμικότητα, ε, και στη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό, αυτή η προστασία βεβαίως έχει ως στόχο να ωφελήσει τους δημιουργούς αλλά και τους χρήστες. Τα τελευταία χρόνια οι παραβιάσεις αλλά και οι παραχαράξεις και παραποίησεις όπως και περιπτώσεις πειρατείας έχουν αυξηθεί αστρονομικά και ιδίως με τη χρήση του διαδικτύου. Εκεί γίνεται μεγάλη ε, παραποίηση των δικαιωμάτων και παραβίαση των διεθνών κανόνων. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη για να ενισχύσουν την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων με την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου παραποίησης και πειρατείας προσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ε, υπό την εποπτεία της Κομισιόν βεβαίως. Το παρατηρητήριο αυτό βέβαια αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Όχι μόνο διότι πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, αλλά θα πρέπει και να λειτουργήσει αποδοτικά. Εδώ η Κομισιόν προτείνει, λοιπόν, και εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση, το παρατηρητήριο να λειτουργεί με ε, μια βέλτιστη σχέση κόστους κόστους-οφέλους και να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εξοικονόμηση κλίμακας και ε, δαπανών, κόστους. 40.000 ευρώ λοιπόν μπορούν να εξοικονομηθούν από τον προϋπολογισμό διότι το κόστος ε, τη λειτουργίας του παρατηρητηρίου θα εποπτεύονται από το, την, ε, το, το πλαίσιο εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς, από το γραφείο εναρμόνισης. Βεβαίως τα διανοητικά δικαιώματα άπτονται και πολιτιστικών θεμάτων και θα πρέπει να φροντίσουμε, να εξασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε την αηφόρο προστασία και ανάπτυξη των ε, πολιτιστικών διανοητικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό ζητούμε, ε, δεδομένου ότι παραβιάσεις, παραποιήσεις και πειρατείες έχουν αυξηθεί και δει στο διαδίκτυο, το παρατηρητήριο θα πρέπει να παρακολουθεί σήματα αλλά και αντιγραφές. αντιγραφές θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι συνεδριάσεις του παρατηρητηρίου θα γίνονται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και θα πρέπει ε, στο παρατηρητήριο να συμμετέχουν και πολιτιστικοί φορείς. Όχι μόνο εκπρόσωποι ε, της βιομηχανίας, ε, του οικονομικού φορέα, νομικών εκπροσώπων, αλλά και πολιτιστικοί φορείς και οι το παρατηρητήριο θα λειτουργεί ε, προσφέροντας υπηρεσίες πληροφόρησης, ε, υλικό ευαισθητοποίησης και ε, επίκαιρο υλικό για τις, με πληροφορίες κλπ. και θα απαντά σε ερωτήματα που αφορούν την παραβίαση διανοητικών δικαιωμάτων. Το παρατηρητήριο επίσης αυτό δεν θα πρέπει να ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα, όπως το προβλέπει η Κομισιόν, διότι δεν, ε, αυτό ξεπερνάει τις αρμοδιότητες ενός τέτοιου φορέα, το οργανωμένο έγκλημα. Δεν θα ασχολείται λοιπόν με τέτοιου είδους παραβιάσεις και παραποιήσεις. Ε, ούτε επίσης θα κάνει μία αξιολογήσεις ε, οργανωμένων εγκληματικών ενεργειών στο θέμα της παραποίησης και της πειρατείας ε, στα οποία δεν θα μπορέσει να ε, ανταποκριθεί. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι πολλά από τα πειρατικά προϊόντα, τα προϊόντα μαϊμούδες, όπως λέμε, βασίζονται στην αντιγραφή γνωστών επώνυμων προϊόντων, αλλά πιστεύω ότι η παρακολούθηση αυτού του τεράστιου θέματος σε διεθνές επίπεδο θα ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του παρατηρητηρίου. Ε, ε καταρχάς θα πρέπει το παρατηρητήριο αυτό, όπως, όπως σας είπα, να λειτουργεί στο πλαίσιο εναρμόνισης της ερωτηρικής αγοράς, ε, να κάνει εξοικονόμηση κόστους και κλίμακας και αν έχετε ερωτήσεις παρακαλώ να μου τις θέσετε. Ε, ευχαριστώ Σαμπίνα, η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς την εισηγήτρια. Και εγώ πιστεύω ότι η ενσωμάτωση του παρατηρητήριου υπό το γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς είναι μια πάρα πολύ λογική διαδικασία και θα του επιτρέψει να λειτουργήσει με ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πιο αποδοτικά θα παρακολουθεί τις παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και θα έχει και τη δυνατότητα καταπολέμησης αυτού του φαινομένου που όλα αυξάνεται θα έχω μία-δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, διευκρινιστικές μάλλον, στις τροπολογίες. Τροπολογία 7... Ε, αναφέρονται οι λέξεις της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής. είναι μια διαφορετική έννοια αυτή, ε, από αυτή που χρησιμοποίησε καταρχάς η Κομισιόν, η οποία αναφέρεται στην καταπολέμηση της ε, παραποίησης και σπηρετής συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού. Γιατί προσετέθη αυτό το μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Εν συνεχεία, ε, η τροπολογία η οποία αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών εννοεί συλλογή πληροφοριών για συλλέγει πληροφορίες για να γίνει μια καλύτερη ανάλυση της κατάστασης στην αγορά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πληροφορίες για αποθήκευση, ε, ένα είδος ε, τράπεζα πληροφοριών. Και τροπολογία 11 που προβλέπει μια δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα κλπ. κλπ, κλπ που θα προσφέρει πληροφορίε, ενημέρωση, αλλά μήπως υπάρχει ο κίνδυνος αν το δεχτούμε αυτό με τόσες λεπτομέρειες ότι το παρατηρητήριο θα προσφέρει πληροφορίες στους πειρατές. Δηλαδή θα δίνει τόσες πολλές πληροφορίες και σε τόσες λεπτομέρειες που θα διευκολύνει το έργο των παραχαρακτών και των πειρατών. Ε, μήπως λοιπόν σε αυτή την 11 θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τι εννοούμε με αυτήν την ε, δημόσια προσβάσιμη πλατφόρμα. Ε, κατά τα άλλα, η αναφορά και του πολιτιστικού τομέα, των καινοτομιών, του design, όλα αυτά και αυτά θα πρέπει να τα καλύψει βέβαια στο παρατηρητήριο, στο έργο του, σε εργασίες του. Η Μαρία Κουτσέτ. Ευχαριστώ. Εμένα μου δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες το γεγονός ότι το παρατηρητήριο θα περάσει στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς. Καταλαβαίνω ότι για λόγους εξοικονόμησης θα ήταν καλό, όμως μου δημιουργεί ανησυχίες γιατί στην ουσία διαχέουμε και απαλύνουμε τον τομέα αυτό, τον τομέα του πολιτισμού. Μιλάμε για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία αλλά και να υπάρχει πρόσβαση και προσβασιμότητα σε θέματα πολιτισμού. Το γεγονός όμως ότι καταργείται το παρατηρητήριο και περνά στην εσωτερική αγορά σημαίνει ότι ξεχνάμε, διαχέουμε κάθε δυνατότητα ιδιαιτερότητας και το πολιτιστικό δεν το βλέπουμε σαν θέμα ιδιαιτεροτήτων που θα μπορούσαμε ούτε προβάλλουμε το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην προσβασιμότητα στην ε, πληροφόρηση. Δεν έχουμε και την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και η Σαμπίν εργάστηκε με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα όμως να το δούμε λίγο πιο ήρεμα, γιατί εμένα μου προκαλεί μεγάλες ανησυχίες αυτός ο μετασχηματισμός. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την κυρία Φεράιν για τις, ε, την εισήγησή της. Εγώ θα πω κάτι βασικό και γι' αυτό θα επικρίνω την πρόταση της Κομισιόν σε δύο σημεία. Διότι λείπει η βασική ισορροπία μεταξύ των δημιουργών και δικαιούχο προστασίας και από, από την άλλη μεταξύ των δικαιούχων των δικαιωμάτων, δηλαδή οι δημιουργοί και οι εκτελεστές, αν θέλετε. Προσωπικά, ε, κάπως ανησυχώ όταν, μιλά, όταν αναφέρονται σε τεχνικά συστήματα, σε συστήματα περίπλοκης ε, τεχνολογίας. Ξέρουμε τις συζητήσεις που γίνονται και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα, για, το δικαιώμα... για τα δικαιώματα αυτά, τα διανοητικά δικαιώματα και κατά πόσον οι πάροχοι, οι providers είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν προφορίες για το πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οι χρήστες οι πάροχοι διαδικτυακών δηλαδή υπηρεσιών αν ε, θα πρέπει να δίνουν ή να μην δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οι χρήστες τους ε, και για το τι ε, ακριβώς χρησιμοποιούν, ποιες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν. Βλέπετε λοιπόν μία μεγάλη μάχη που γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ πάροχων υπηρεσιών, παρόχων ε, υπηρεσιών διαδικτύου και χρηστών. Πρέπει λοιπόν από τη μία πλευρά να προστατεύσουμε το δικαίωμα των δημιουργών και από την άλλη όμως και τα δικαιώματα των χρηστών. Δεν είναι δυνατόν να, να δημιουργήσουμε μία υποδομή αυστηρή και η οποία θα εμποδίσει την ελεύθερη ροή ε, διανοητικής εργασίας, διανοητικών προϊόντων μέσα στο οποία βεβαίως εννοώ και, τα, και το διαδίκτυο, τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Όπως και να το κάνουμε υπάρχουν δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά υπάρχει ε, τα downloads που κάνουμε όλοι μας στο σπίτι μας. Ε, κατεβάζουμε ένα-δύο ε, τραγούδια, πληροφο... κάνα βίντεο ή κάποια εκπομπή για ιδιωτική χρήση. Και από την άλλη υπάρχουν φορείς ή άτομα τα οποία κατεβάζουν εκατομμύρια, χιλιάδες τραγούδια και έτσι κλέβουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τους δημιουργούς. Λοιπόν, ε, υπάρχει και η σχετικότητα χρήσης, έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα θεμελιώδες ε, ζήτημα το οποίο αφορά τον τρόπο χρήσης. Αλλά η κυρία Πακ, η κλεψιά είναι κλεψιά. Τώρα, εάν κλέβεις μία καραμέλα ή μία ολόκληρη τούρτα, τι μέγεθος έχει το κομμάτι που κλέβεις, μα δεν συζητάμε αυτό. Ο κλέφτης είναι κλέφτης. Η κυρία Χίπνερ, ευχαριστώ Ντόρις. Ε, συνεχίζω μετά αυτά που είπε η Εύα ε, Είναι γεγονός ότι υπήρχαν παράνομες πλατφόρμες μέχρι τώρα οι οποίες με περιεχόμενο από τρίτους δημιουργούς ε, εξασφάλιζαν κέρδη χωρίς να ανταμείψουν ή να καταβάλουν τα δικαιώματα στους δημιουργούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία ένας ε, πάροχος, προμηθευτής ε, κινηματογραφικών έργων μέσω του διαδικτύου, ε, διαμέσου του οποίου μπορείς να κατεβάσεις μία ταινία χωρίς να πληρώσεις κανένα δικαίωμα. δικαίωμα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να επιτρέψουμε ένα τέτοιο επιχειρησιακό μοντέλο, ένα τέτοιο business model, το οποίο να υπονομεύει το δικαίωμα δίκαιης, ε, δίκαιου κέρδους των δημιουργών μια ταινίας ή ενός μουσικού έργου. Το επόμενο ερώτημα, που είναι πάρα πολύ ε, καυτό. Οι νέοι, οι νέοι, οι νέοι άνθρωποι κάνουν το εξή. Ε, πράγματα τα οποία έχουν αγοράσει, θέλουν να τα μοιραστούν με άλλους, ε, ε, αγοράζουν ένα CD ας πούμε, την κοπιά, κοπιάρει το CD και το χαρίζει σε 5-6 φίλους του. αυτό έχει ρυθμιστεί, θεωρείται προσωπικό δώρο. Αλλά στον ψηφιακό κόσμο τα πράγματα έχουν γίνει διαφορετικά. Υπάρχει μία ε, κοινή ε, απόκτηση, ε, μοιράζονται δηλαδή εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ένα κοινό πνευματικό υλικό, ένα υλικό με διανοητικά δικαιώματα του δημιουργού. Δεν λέω ότι πρέπει να περιορίσουμε την ροή των πολιτιστικών προϊόντων, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε τον ασέμητο αυτό ανταγωνισμό μέσω διαδικτύου και την υφαρπαγή των νόμιμων δικαιωμάτων από εκατομμύρια χρήστες. Πρέπει λοιπόν να, να αναρωτηθούμε το εξής. Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε τις μη εξουσιοδοτημένες αντιγραφές ε, από τις εξουσιοδοτημένες αντιγραφές. Εάν είναι εξουσιοδοτημένη η αντιγραφή θα πρέπει κάποιος να πληρώσει. Οπότε υπάρχει ένα ξεκάθαρο επιχειρησιακό μοντέλο, θέλεις να κατεβάσεις κάτι στον κομπιούτερ σου ή να το αντιγράψεις, πληρώνεις ε, και είσαι ωραίος και νόμιμος. Αλλά όταν έκλεισε ας πούμε το Napster παλιά δημιουργήθηκε το Καζά, μετά το Καζά δημιουργήθηκε το Spotify. Το Spotify στην αρχή ήταν δωρεάν, τώρα όμως πρέπει να πληρώσεις για να μπορέσει να ακούσεις τη μουσική βιβλιοθήκη. Αυτό το είναι αυτή η νομοθεσία χειρίζεται με μεγάλη σοβαρότητα τα δικαιώματα των δημιουργών αλλά και, να, και σέβεται παράλληλα τα δικαιώματα των χρηστών. Πρέπει να βρούμε μία σωστή ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Είναι δύσκολο έργο αυτό το να βρούμε μια σωστή υπηρεσία χωρίς να ε, παραβιάσουμε θεμελιώδη δικαιώματα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό θα πρέπει το παράνομο υλικό ή το υλικό του οποίου γίνεται εμπορία παράνομα να μην το επιτρέψουμε. Και επίσης πρέπει να ε, συμφωνήσουμε στην ορολογία. Τι θα πει ιδιωτικό δίκτυο, ποιο είναι ιδιωτικό δίκτυο, ηλεκτρονικό δηλαδή και ποιο δεν είναι. Ε, αν θέλουμε να αναπτύξουμε την ψηφιακή αγορά, βεβαίως το πράγμα το οποίο θέλουμε, ε, δεν θα πρέπει να περιορίσουμε <clears throat> τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης. Όμως, ταυτόχρονα, πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα διανοητικά δικαιώματα. Ας μην ξεχνάμε ότι καθημερινά δημιουργούνται νέα, νέες ιστοσελίδες, νέα sites από τα οποία μπορεί κανείς παράνομα να κατεβάσει πολιτιστικά προϊόντα. Και εγώ πιστεύω ότι η έκθεση της Κομισιόν ε, ή αυτά που είπε ο Ζήκρβιτ Κάουντα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, η αυτα που ειπε ο ζηκρβιτ προσφέρει στην επιτροπη εσωτερικης αγορας η εκθεση της Κομισιόν δεν προσφέρει την ιδανική λύση και θα πρέπει η Σαμπίν να εκφράσει την γνώμη της απερίφραστα ε, και να προσπαθήσει να διευκρινίσει, να ζητήσει δηλαδή να διευκρινιστεί τι είναι δημόσιο αγαθό και τι είναι ιδιωτικό. Ε, ε, εξουσιοδοτημένη αντιγραφή μπορεί να την δεχτούμε. Μη εξουσιοδοτημένη είναι παράνομη και κλεψιμέα. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Η Σαμπίνα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η πρόταση της Κομισιόν δεν στοχεύει στη νέα ρύθμιση για την προστασία του copyright. Εδώ πρόκειται για μια μετατόπιση αρμοδιοτήτων, ούτε καν μετατόπιση, αλλά μια νέα διάρθρωση ε, μιας υπηρεσίας που ήδη υπάρχει και ανάθεση νέων καθηκόντων. ανάθεση μάλλον ορισμένων καθηκόντων που έχουν σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία. Εδώ δεν πρόκειται για μια νέα νομοθεσία, νέους κανόνες για το copyright. Αν χρειαστεί αργότερα να αλλάξουμε το copyright και όλη τη συναφή νομοθεσία θα γίνει, αλλά σε άλλο επίπεδο. Αυτό που εννοώ με την τροπολογία 7 και οι περισσότερες παρατηρήσεις προέρχονται από γερμανούς συναδέλφους. Unauthorized copies, λέει, ε, στα, γερμανικά, ε, στα αγγλικά. Εγώ έχω μόνο το γερμανικό κείμενο και δεν νομίζω ότι είναι ακριβή η μετάφραση, επειδή η μετάφραση έγινε με μεγάλη ε, χρονική πίεση. δουλέψαμε καταρχάς στο αγγλικό κείμενο, εν συνεχεία μεταφράστηκε στα γερμανικά και στις άλλες γλώσσες. Το αρχικό κείμενο ήταν το αγγλικό. unauthorized non-authorized copies, unauthorized copies, μη ε, εξουσιοδοτημένες αντιγραφές. Ε, μπορούμε να βάλουμε και τη λέξη commercial copies, ε, unauthorized commercial copies. Μπορούμε να συμπληρώσουμε έτσι τον ορισμό, μαζί με το counterfeiting και το piracy, την παραποίηση και την πειρατεία. Να προσθέσουμε και τις μη εξουσιοδοτημένες κόπιες απομιμήσεις ή αντιγραφές, αν θέλετε, ανάλογα με τη μετάφραση. Ε, ακριβώς αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε ακριβώς την υπερβολική χρήση αυτών των, αντι, των ε, αντιγραφών που γίνεται σε ιδιωτικό χώρο, σε ιδιωτικό επίπεδο, συνεχεία γίνεται εμπορική εκμετάλλευση. Ε, και πάλι επανέρχομαι στο θέμα της συμμετοχής των πολιτιστικών φορέων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν επικεντρωνόταν υπερβολικά πολύ στα οικονομικά συμφέροντα ε, της, ε, των διάφορων κλάδων ε, που, που, που άπτονται αυτού του θέματος και όχι τόσο πολύ με τους πολιτιστικούς φορείς. Γι' αυτό ζητώ το παρατηρητήριο, στο παρατηρητήριο να συμμετέχουν και να εκφράζουν την άποψή τους και πολιτιστικοί φορείς. Έτσι ώστε στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτού του παρατηρίου να ακούγεται περισσότερο και πιο έντονη η, η, η πλευρά των, του πολιτισμού, των πολιτιστικών ε, αρμοδίων. Το παρατηρητήριο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα αυτή την πτυχή του copyright. διότι περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην αγορά των ε, ε, πολιτιστικών προϊόντων. Όχι τόσο πολύ ε, τα δικαιώματα προϊόντων βιομηχανικών ή άλλων αγαθών και εμπορευμάτων. Μας ενδιαφέρει η διανοητική ιδιοκτησία καλλιτεχνικών πολιτιστικών προγραμμάτων. Ναι, σωστά αυτή η έκθεση αναφέρεται στο παρατηρητήριο. αυτό είναι το, ο στόχος. Και αναρωτιέμαι εάν με αυτή την οδηγία προκαταλαμβάνουμε το δεύτερο στάδιο ε, αντί να μελετήσουμε το πρώτο στάδιο. Προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Μήπως δηλαδή προτρέχουμε εμείς θέλουμε να επιβληθεί μια λογική ισορροπία. Σωστό. Αλλά αυτές οι ιδιωτικές αντιγραφές που γίνονται ε, και με το παρελθόν που είχαμε όσον αφορά την αναλογική τεχνολογία έναντι της ψηφιακής σήμερα. Μήπως πρέπει να διευκρινίσουμε πρώτα όλα αυτά τα θέματα ορολογίας, οριοθετήσεις τομέων, πριν προχωρήσουμε σε πιο περίπλοκα. Η Κομισιόν θα μας φωτίσει, θα μας απαντήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε καταρχάς την έκθεση, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας για το ζήτημα αυτό. Ήδη εξ αρχής θεωρούσαμε ότι το ευρωπαϊκό αυτό παρατηρητήριο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους πολιτιστικούς φορείς. Επομένως, ε, είμαστε σαφώς υπέρ του να υπάρχει μια διευκρίνηση για το ζήτημα αυτό μέσω τροπολογίας. Όσον αφορά τώρα τους λόγου λόγους για τους οποίους θα πρέπει το παρατηρητήριο να περάσει στο γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, πρέπει και εμείς να πούμε, όπως είπε και η εισηγήτρια ότι θα υπάρχει μια καλύτερη υποδομή, καλύτερη χρηματοδοτική πόρη, καθώς επίσης και ένα προσωπικό το οποίο θα είναι εξειδικευμένο στο ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συλλέξουμε και πιο χρήσιμες πληροφορίες, γιατί αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος. Δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε περαιτέρω, δεν θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις, θέλουμε να συλλέξουμε καλύτερες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στο μέλλον τους συνομοθέτες για τα ζητήματα αυτά τα οποία συζητάμε ακόμα και σήμερα. Καταλαβαίνω λοιπόν τις ευαισθησίες που έχουν εκφραστεί όσον αφορά τον εντοπισμό των περιπτώσεων απομίμησης και αντιγραφής. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως να δούμε αν θα γίνει αυτό με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει μόνο για τον έναν ή τον άλλον τομέα. Δεύτερον, τα μέλη του παρατηρητηρίου, η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό αυτό παρατηρητήριο και η καλύτερη εκπροσώπηση, όπως είπατε, του πολιτιστικού τομέου, τομέα, με συγχωρείτε, δεν είναι παγιωμένη, δεν είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Προφανώς η συμμετοχή μπορεί να είναι πιο ανοιχτή, πιο δυναμική. Και όσον αφορά τώρα τους εκπροσώπους του εμπορικού ή του ιδιωτικού τομέα, η συμμετοχή τους θα εξαρτηθεί από τον τομέα που κάθε φορά εξετάζουμε. Αν, για παράδειγμα, το ζήτημά μας είναι η πειρατεία, τότε προφανώς στο παρατηρητήριο θα πρέπει να συμμετέχουν και μέλη τα οποία εκπροσωπούν τον, τους τομείς που πλήττονται από την πειρατεία. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα παρατηρητήριο πολύ πιο αποτελεσματικό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παρατηρητήριο το οποίο έχει απλώς μια γραμματεία και πολύ περιορισμένους πόρους. Επίσης, στο, στο παρατηρητήριο προτείνουμε να υπάρχουν και εκπρόσωποι παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εργασία που θα γίνει, αλλά και για τη διασύνδεση του παρατηρητήριου με τους νομοθέτες και συνομοθέτες. Μπορείτε κατά αυτόν τον τρόπο να καθορίσετε και εσείς τις προτεραιότητες εργασίας του παρατηρητηρίου και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω βέβαια και σε περαιτέρω ερωτήσεις. Όσον αφορά την μη εξισοδοτημένη αντιγραφή και ξέρω ότι αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε σχέση με τον όρο πειρατεία. Είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να καλυφθούν τα πάντα μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο όμω η εισηγήτρια αποφάσισε να προσθέσει και τον όρο μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Ουσιαστικά θέλησε να δώσει μια πιο σαφή χρειά και να μην χρησιμοποιείται μόνο όρο όρος πειρατεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, λέει η κυρία Πακ, δεν απαντήσατε στο ερώτημα των δύο κυρι... κυρίων, κυριών. Γιατί ε, κάνετε αυτό το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο. Γιατί δεν περιμένουμε πρώτα την ε, υιοθέτηση της οδηγίας για το copyright και εν συνεχεία να κάνουμε την μετάθεση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Για ποιο λόγο το παρουσιάζετε αυτό τώρα. Κοιτάξτε, αν δούμε τα πράγματα από χρονολογική σειρά, το παρατηρητήριο ήδη υπήρχε και λειτουργούσε. Και η πρόταση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια μέρα με τη στρατηγική που έχουμε για τα πνευματικά δικαιώματα και εκεί πέρα προβλέπονται και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες και για τον τομέα του copyright που προφανώς θα σας απασχολήσουν. Κατά την άποψή μας λοιπόν θεωρούμε ότι δεν έχουμε ξεκινήσει ανάποδα. Είναι ένα παρατηρητήριο το οποίο ήδη υπάρχει και έχει σε άλλες συζητήσεις που είχαμε. Ορισμένοι είπαν ότι το παρατηρητήριο θα μπορούσε να ασχολείται και με κάποια άλλα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε πάντως ότι το παρατηρητήριο θα μπορούσε να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα όταν αποφασίζουν για ζητήματα όπως η προστασία δημοτικών δικαιωμάτων, η πειρατεία κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες όμως για το πώς επιβάλλονται οι σχετικές νομοθεσίες στα κράτη-μέλη, για το πώς αποδοτικά είναι τα συστήματα αυτά. Έτσι λοιπόν μέσω του παρατηρητηρίου θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς στη συνέχεια να βελτιώσουμε την προτινόμενη νομοθεσία. Αυτή την εξήγηση μπορώ να σας δώσω. Once πάλι το λόγο. Ναι, και εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν, προκαταλαμβάνουμε νομοθετικές προτάσεις ε, ή τρόφου, τρόπους με τους οποίους θα ελέγξουμε διάφορα ζητήματα. Το θέμα είναι, όπως είπε και η Επιτροπή, ότι υπάρχει ήδη ένα παρατηρητήριο με οργανωτικές δομές, αλλά οι δομές αυτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, σωστά στο έργο του παρατηρητηρίου εάν δεν καλυφθεί από το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς εάν δημιουργήσουμε αυτή τη συνέργεια θα, επιτύχουμε, θα επιτύχει το παρατηρητήριο με καλύτερη συλλογή πληροφοριών, καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση για παράνομες δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα ε, στον οποίο έχει αρμοδιότητες. Και αυτό είναι και ο στόχος του παρατηρητηρίου. Δεν προκαταλαμβάνουμε μελλοντικέ ρυθμίσεις, δεν προκαταλαμβάνουμε ε, μελλοντικά μέτρα για το copyright. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αποφασίσουμε μέσω του παρατηρητηρίου αν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε ορισμένου τομείς ή όχι. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στον φορέα αυτό να κάνει τις σωστές αναλύσεις βάσει των σωστών πληροφοριών που θα συλλέγει. Α, δεν θα πρέπει ε, επίσης το, να ζητήσουμε από το παρατηρητήριο να, να εκτελεί και έρευνες, research που μπήκε κατά λάθο στο κείμενο, συλλογή πληροφοριών, ε, information, όχι research. Μην το αναφέρσουμε και επιστημονικές εργασίες. Α, ωραία, λέει η, η κυρία Πακ. Ε, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Προθεσμία τροπολογιών 13 Οκτωβρίου, την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα σύστημα, έτσι, ε, σεβασμού της προθεσμίας των τροπολογιών. 12 το μεσημέρι, 13 Οκτωβρίου, τέρμα. Και θα ψηφίσουμε στις 10 Νοεμβρίου. Και αρμόδια επιτροπή θα ψηφίσει ολόκληρη την έκθεση τον Δεκέμβριο. Η επί, η επί επιτροπή. Σημείο 6. επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Δίνω και πάλι το λόγο στη Σαμπίνετολ το ε, Βερχάιεν. Λοιπόν, ε, εδώ έχουμε μία συζήτηση επί της ουσίας και όχι επί των τύπων ποιος ε, θα παρατηρεί τι, πού, πώς και γιατί. Ε, το θέμα είναι πώς θα χειριστούμε αυτό το μεγάλο όγκο ορφανών έργων της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς μας, του πολιτισμού της Ευρώπης, που, στα οποία έχουμε πρόσβαση. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μία πρόταση για ε, οδηγία για την κάλυψη όλων αυτών των ορφανών έργων, βιβλίων, κειμένων κλπ. Ε, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει ένας πλήρης κατάλογος ταυτοποίησης αυτών των έργων. Ε, πρέπει να, να δημιουργηθεί ένα αρχείο. Ναι, η κυρία Πακ διακόπτει, διότι ομιλείται μιλά με ταχύτητα φωτό και εμεί καημένοι διερμηνεί δεν, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Προσπαθεί να την ε, να μιλήσει πιο σιγά. Λοιπόν, 500 ε, εκατομμύρια κάτοικοι εποφελούνται από αυτά τα έργα και είναι πολύ καλό να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα έργα, πνευματικά έργα με την ψηφιοποίηση και την αρχαιοθέτηση αυτών των ερφανών έργων θα συμπληρώσουμε ένα μεγάλο κενό στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Ε, πάρα πολλά ορφανά έργα αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε ραδιοφωνικές βιβλιοθήκες, σε αρχεία, ε, σε κινηματογραφικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες ταινιών, ταινιοθήκες συγγνώμη κλπ. Και γι' αυτό η οδηγία αυτή έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα μιας διασυνοριακής χρήσης αυτών των έργων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν ορφανά έργα όταν δεν έχει ανεβρηθεί ο δημιουργός, ο δικαιούχος και έτσι θα συμβάλλουμε στην ε, πολυπολιτισμική διάσταση της Ευρώπης. Ιδιαίτερα ε, στο, στα τυπωμένα ε, κείμενα, περιοδικά, βιβλία... Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ορθανές εκδόσεις. Πολλές κυβερνήσεις κρατών μαλλών έχουν ξεκινήσει αυτή την ψηφιοποίηση των αρχείων και αυτή η οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα ε, μιας ε, σωστής αποθήκευσης και διευκόλυνσης στη χρήση των ενδιαφερομένων των έργων αυτών. Είτε είναι ραδιοφωνικές εκπομπές, είτε είναι ντοκιμοντέρ, είτε είναι ταινίες, είτε είναι τυπωμένα προϊόντα, βιβλία και περιοδικά. Ε, πάρα πολλά τέτοια πνευματικά έργα δεν χρησιμοποιούνται διότι δεν ξέρει κανείς αν μπορούν να διατεθούν ή όχι. Ε, θα πρέπει λοιπόν η οδηγία να έχει την κατάλληλη διατύπωση και να λέει ότι ε, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η χρήση ε, ενός ε, ε, προϊόντος, ενός έργου, όταν δεν μπορούμε να βρούμε τον αρχικό δημιουργό, παραδείγματος χάρη, μιας φωτογραφίας. Ας πούμε ότι είναι ένα βιβλίο και σε μια φωτογραφία δεν μπορούμε να βρούμε από κανένα αρχείο ποιος την τράβηξε. Δεν είναι τότε λοιπόν σωστό να απαγορεύσουμε πλήρως τη χρήση αυτού του βιβλίου, τη διανομή αυτού του βιβλίου πρέπει πριν ε, ε, διαπιστώσουμε ότι ένα έργο είναι ορφανό και ότι έτσι θα επιτρέψουμε τη χρήση του, να γίνει μια σωστή έρευνα ε, και μια μεγάλη προσπάθεια, σωστή προσπάθεια να βρεθεί ο δικαιούχος αν υπάρχει των διανοητικών δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να απευθυνθούμε σε συλλεκτικές οργανώσεις, σε συλλέκτες, ε, που μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα, διότι ε, οι συλλέκτες και συλλεκτικές ενώσεις, φορείς ε, έχουν πολλές πληροφορίες για δημιουργούς πνευματικών έργων και επίσης και πάλι πρέπει να αποτανθούμε σε πνευματικά ιδρύματα, ε, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και να τους βοηθήσουμε εάν θέλουν να διαθέσουν υλικό και δεν μπορούν να κάνουν όλη την έρευνα να τους βοηθήσουμε στην ε, χρησιμοποίηση αυτού του υλικού. Ε, αυτές είναι οι βασικές ιδέες για τις χρήσεις που θέλουμε να επιτρέψουμε στα ορφανά έργα μπορεί να παρέβλεψα. Μερικά είναι και μερικά έργα τα οποία είναι ημιορφανά, δηλαδή εν μέρη έχουμε, έχουμε βρεθεί οι δικαιούχοι, αλλά όχι όλοι. Αυτά τα βασικά σημεία της πρότασης. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα σε αυτό το θέμα και όσον αφορά τις τροπές απολογίες θέλω να πω το εξή. Η πρόταση της Κομισιόν, η αρχική της πρόθεση είναι πάρα πολύ σωστή. Πρέπει να βρούμε μια λογική, ε, μια ευλογή ε, διαδικασία να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έργα. Έτσι δεν είναι. Ε, χωρίς να μπλέξουμε σε νομικά ζητήματα κλασικά λογοτεχνικά έργα παραδείγματος χάρη ε, όπου έχουν απελευθερωθεί δεν υπάρχει πλέον διανοητικά δικαιώματα εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ σωστή χρήση των δικαιωμάτων αυτών ε, αυτό σε ένα βιβλίο αλλά σε ένα οπτικοακουστικό θέμα εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί από, διαφορετικούς, ε, από διαφορετικές ειδικότητες ρώτησα ε, τι σημαίνει αυτή αυτή η ανέβρεση των δημιουργών. 1,3 εκατομμύρια ε, τηλεοπτικά προγράμματα, διότι ρώτησε την, ένα γερμανικό κανάλι, 1,3 εκατομμύρια τηλεοπτικά προγράμματα παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Ε, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει η διευκρίνηση εάν μία τηλεοπτική εκπομπή είναι ορφανή ή όχι. Και αυτό μόνο για ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε, αν κάποιος θέλει να ε, διαπιστώσει και να ελέγξει εάν υπάρχουν ορφανά τηλεοπτικά έργα ή ορφανές τηλεοπτικές εκπομπές θα πρέπει να αναφερθεί σε εκατομμύρια εκπομπές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Α, αυτή λοιπόν η έρευνα που εχουν γινει κατα τη διαρκεια των τελευταιων δεκαετιων αυτη λοιπον η ερευνα που απαιτειται για τα οπτικοακουστικά προϊόντα, οπτικοακουστικά έργα δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εφαρμόσιμη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε λογικοί και όσον αφορά τα οπτικοακουστικά θεάματα ή έργα χρειαζόμαστε ένα απλούστερο μοντέλο. Όπως ας πούμε το Extended Collective Licensing System, δηλαδή ένα διευρυμένο σύστημα παροχής αδειών εκμετάλλευσης, ε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προϊόντα και για να μπορεί κάποιος να έχει γρήγορη πρόσβαση σε ένα αρχείο και να πάρει το προϊόν που θέλει να χρησιμοποιήσει και όχι να χρειαστεί να κάνει μία επίπονη και, και μη ρεαλιστική έρευνα των αρχικών δημιουργών και εάν υποθέσουμε ότι κάποιος τελικά ε, παρουσιάζεται και γύρει απαιτήσει ε, διανοητικών δικαιωμάτων. Εάν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό το άτομο ή αυτός ο φορέας να λάβει την αμοιβή που δικαιούται. Εάν λοιπόν ε, κάποιος έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός τέτοιου έργου, δικαιούται τα διανοητικά του δικαιώματα εφόσον μπορεί να το αποδείξει. Αλλά ε, να μην ε, κολλήσουμε με, με, ψήλους, να μην γυρεύουμε ψήλους τάχυρα, να προσπαθήσουμε να βασιστούμε σε μια λογική προσέγγιση και απλή προσέγγιση που να δώσει χρήση στα εκατομμύρια αυτά των προϊόντων. Κύριε Παγιαδέλη ερώτηση δεν έχω νομίζω καταλάβει αν ορφανά είναι μόνο αυτά των οποίων δεν γνωρίζουμε το 100% των κατόχων δικαιωμάτων του ή αν είναι και εκείνο των οποίων έχει λήξει η αν ειναι και εκεινο τον οποιο εχει ληξει η περιοδος ε, των 50 ετών αν θυμάμαι καλά για την οποία, μετά από την οποία ένα έργο είναι ελεύθερο. Επομένω, μια ερώτηση είναι αυτή, δεν ξέρω αν γίνεται σαφής η διατύπωση στο κείμενο των, της, της Επιτροπής Νομικών. Το άλλο ερώτημα είναι αν ε, μπορούμε πάντοτε με σαφήνεια να καθορίσουμε τον, ε, τον κάτοχο ή τους κατόχους. Για παράδειγμα, μία φωτογραφία για την οποία κάποιος πληρώθηκε. Είναι ξεκάθαρο σε, όλη, σε όλα τα ευρωπαϊκά, μέλη τα ευρωπαϊκά κράτη από την ομοθεσία τους ότι ανήκει στον φωτογράφο, στον δημιουργό ή στο περιοδικό ή την εφημερίδα που την αγόρασε αν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα και υπάρχει μια γενικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των δύο αυτών βασικών όρων, ορφανό έργο, κάτοχος δικαιωμάτων, από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Έχω την αίσθηση όμως ότι και συμμερίζομαι τις ανησυχίες της ε, συναδέλφου ότι αν δεν αποσαφηνίσουμε τους όρους θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε ή να κατέληξουμε σε ένα τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, κυρία Σάλκ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, βλέπω ότι γίνεται μία συνεχής αλλαγή στη διατύπωση. Από το καθιστούμε διαθέσιμο, λέμε επικοινωνούμε στη συνέχεια Ενδεχομένω να υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφραση εδώ πέρα ή ουσιαστικά αλλάζει και η ουσία. Για ποιο λόγο γίνεται συνεχώς αυτή η αλλαγή από το making available communicate στο αγγλικό κείμενο. Η ομιλήτρια αναφέρει επίση την αλλαγή διατύπωση στα Ολλανδικά. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάποια πολύ παλαιά έργα τα οποία δεν έχουν ψηφιοποιηθεί δεν είναι περιορισμένα, αλλά είναι διαθέσιμα για το κοινό. Πώς το εξασφαλίζουμε αυτό. Τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό οι ιδιώτες, ο ιδιωτικός τομέας. Πώς μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τρύπελ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό την Ειδική Επιτροπή η οποία μας είχε πει ότι θα πρέπει να βρούμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση και στα στην διευθέτηση της, α, στο, Ευρωπαϊκό, α, στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης έγινε η εκδίκαση μιας, ε, μιας ειδικής περίπτωσης ε, η οποία έθιξε ακριβώς αυτό το θέμα. Μην ξεχνάτε λοιπόν ε, το, το ιστορικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης, το υπόβαθρο. πιστεύω ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει να γίνει μία σωστή έρευνα, μία σχολαστική αναζήτηση. Αλλά εκεί που δεν χρειάζεται ή εκεί που δεν γίνεται, Πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε και πάλι τη σωστή ισορροπία μεταξύ της πληρωμής των πνευματικών δικαιωμάτων και της ε, ε, εύκολης ε, πρόσβασης και της ευκολίας χρήσης των προϊόντων αυτών. Πρέπει να υπάρχουν απλοί μέθοδοι, απλή, απλά μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πολίτης. Γι' αυτό και συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν για τα οπτικοακουστικά προϊόντα. Να χρησιμοποιηθεί αυτή η Extended Collective Licensing, αυτή η συλλογική ε, διαχείριση δηλαδή, η παρατεταμένη συλλογική διαχείριση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πρακτικό τρόπο αυτά τα προϊόντα. Τώρα, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, ότι καταρχάς πρέπει να θεωρήσουμε ως πρωταρχική πηγή το κράτος δημιουργίας. Αλλά εν συνεχεία πρέπει να δούμε όταν παρουσιάζονται δημιουργοί από άλλα μέρη, από άλλες χώρες και όχι τη, τη χώρα όπου δημιουργήθηκε το προϊόν, να λαμβάνονται και αυτονών τα δικαιώματα υπόψη. διότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει κάποιος που συνέβαλε σε αυτή τη δημιουργία και δικαιούται διανοητικά δικαιώματα. Το δεύτερο είναι η συλλογή ε, πληροφοριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, μία σωστή γνώση και ενημέρωση για την κατάσταση των ορφανών έργων, ώστε στο μέλλον να μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε περισσότερα ορφανά έργα, ο στόχος μας είναι να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε στην μελλοντική νομοθεσία να μην υπάρξει, να μην εμφανίζεται πια στο μέλλον. πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα ελέγχθησαν, αλλά δεν ελέγχθη το εξής, ότι υπάρχει, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να δούμε ε, κατά πόσο ένα έργο είναι ορφανό έργο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν έρευνες τεχνική υφή για να το προσδιορίσουμε. Αλλά ποιος θα αναλάβει αυτή την έρευνα, αυτό δεν ελέγχθη και ποιο θα τη χρηματοδοτήσει. Κύριε Πρόεδρε, Πολύ σωστά είπε η συγγήτρια ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τις δικές τους ε, λύσεις και το ίδιο ισχύει για την Φιλανδία και τις βόρειες χώρες. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Στις βόρειες χώρες έχουμε ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται, το παλαιό σύστημα το οποίο μεταξελίσσεται και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με αυτό. Και με βάση αυτό το δεδομένο θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία 15, η οποία είναι πολύ σημαντική για μας. Ίσως φαίνεται μικρή, η οποία βγάζει δύο λέξεις, αλλά σε εμάς αφήνει πολλά περιθώρια να μπορέσουμε να κινηθούμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και θα ήθελα να πω ότι το θέμα των ευρωπαϊκών ε, βιβλιοθήκων είναι δύσκολο μετά την ψηφιοποίηση και μετά την ψηφιοποίησή τους είδαμε ότι θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το έμπλεχο εμπλεκόμενο, εμπλεκόμενο κόστος για να προβούμε σε αυτή την ε, diligent research των συγγραφέων. Μιλάμε για αρχεία, βιβλιοθήκες και ούτω καθεξής. Και εδώ μιλάμε και για ιδιωτικούς φορείς και θα πρέπει να μας το διευκρινίσει η Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει θα προτιμούσα μία εξαίρεση για όλα τα έργα, έργα όμνες, για όλους δηλαδή τους φορείς, έτσι ώστε όταν ιχνηλατηθούν οι συγγραφείς να υπάρχει δυνατότητα αμοιβή. Διότι το κόστος της έρευνας είναι τόσο υψηλό που θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ιχνηλατήσουμε τα ορφανά έργα. Κατά δεύτερον, μιλάμε για συλλογικές αδειοδοτήσεις που είναι μια άλλη μορφή. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί. Εδώ όμως η Επιτροπή έκανε μια επιλογή αρχής και από εκεί και πέρα δεν προχώρησε. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προαπαιτήσεις και πώς έχει η ισορροπία μεταξύ πνευματικών δικαιωμάτων και εξέβρεση συγγραφέων. Διότι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με έργα τα οποία δεν κυκλοφορούν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε ξεχωριστά για τα έργα των βιβλιοθηκών και τα οπτικοακουστικά από την άλλη πλευρά. Ένα άλλο αίτημα είναι να υπάρχει μια τεχνική ουδετερότητα στα πλαίσια της ε, ψηφιοποίησης από τα κράτη-μέλη, να μην υπάρχουν δηλαδή δεσμεύσεις. Και είδα ότι η συνάδελφος προβλέπει η αμοιβή να δοθεί σε συγκεκριμένα πολιτιστικά κέντρα που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ίσως θα έπρεπε κάτι τέτοιο να ισχύει είτε για τις επιχειρήσεις ομαδικών αδειοδοτήσεων είτε για τα Ινστιτούτα ή φορείς που ψηφιοποιούν αυτά τα έργα που αναλαμβάνουν πολύ μεγάλο κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να αμείβεται αυτός ο οποίος διαθέτει στο κοινό αυτά τα έργα. Χρειάζονται λοιπόν αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μιλάμε και για ιδιωτικούς και για δημόσιους φορείς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συνάδελφος Μπερλιγκουέρ. Ευχαριστώ. Εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όπου συζητιέται αυτό το θέμα in primis. Και το λέω αυτό γιατί είτε, είτε σε εκείνη την Επιτροπή είτε εδώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να αμείβουμε τους καλλιτέχνες ή τους συγγραφείς και αυτό δεν γίνεται επαρκώς. Όμως δεν πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία όταν έχουμε να κάνουμε με έργα όπου έχουν αποβιώσει οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς ή δεν τους γνωρίζουμε. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ορισμένες γενικές αρχές, αλλά υπάρχει η αιμονή να αμείγονται ακόμα και οι νεκροί. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και άρα υπάρχει πίεση από τις επιχειρήσεις διαχείρισης του έργου του Φανόντα. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε προσβασιμότητα σε αυτά τα έργα. Πρόκειται για μεγάλες, μεγάλα έργα και πολλά έργα. Γιατί τη στιγμή που ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται για την αμοιβή και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα τους ενδιαφέρε όμως η διάδοση των έργων τους δηλαδή θα θέλαν ψηφιοποίηση. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της έρευνας, της ε, έγκαιρης έρευνας ή της επιταχυμένης έρευνας στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται λόγος για συλλογικά σχήματα επιχειρήσεων. Εδώ όμως ερχόμαστε σε μία σχέση σύγκρουσης, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι η θέση της Επιτροπής θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί αν αρκεστούμε σε αυτά που προτείνει η Κομισιό, δεν θα έχουμε ψηφιοποίηση δεν προτρέπουμε την ψηφιοποίηση, δηλαδή τη μέγιστη διάδοση αυτών των έργων. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι διατάξεις, οι ρυθμίσεις οδηγούν σε υποψίες ότι θέλουμε να βρούμε και αυτούς που δεν υπάρχουν. Ξέρω ότι υπερβάλλω, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η λανθάνουσα πρόθεση. Ευχαριστούμε κύριε Μπερλίνγκουερ. Πολλά από αυτά που είπατε τα συζητήσαμε ήδη στην αρχή τη συζήτηση, αλλά τα επαναλαμβάνουμε. Σαμπίνε, θες να, πα... να μιλήσεις τώρα ή μετά από την Κομισιόν. Θα ήθελα, ε, λέει η μετα απο την κομισιον θα ηθελα λεει σαμπινε να απαντήσω σύντομα. Καταρχάς, οι συλλογικές αυτές ε, ε, εταιρείε ε, είναι μία δυνατότητα, δεν, δεν είναι υποχρεωτικές θα πρέπει ακριβώς να ενεργούν ως ένα ε, δίκτυο προστασίας. Όταν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε ένα έργο, Α, δεν, δεν εννοείται ότι κάποιος ο οποίος ε, ε, είναι ο δημιουργός, είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, έχει αποβιώσει. Μπορεί να ζει ο άνθρωπος ή τέλος πάντων ο φορέας, αλλά ε, ένα τέτοιο copyright κληρονομείται κιόλα. Η πνευματική ιδιοκτησία, το copyright ενός, ε, του, πατέρα, ας πούμε, ή ενός δημιουργού μπορεί να κληρονομηθεί στα παιδιά του και τα παιδιά να αποφεληθούν ή άλλοι κληρονόμοι από τα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, προσπαθούμε να εδραιώσουμε την ευρύτερη δυνατόν προστασία Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι ε, αυτοί που κάνουν την ψηφιοποίηση θα πρέπει να μας προσφέρουν και τις υπηρεσίες για την αναζήτηση των ε, κατόχων δικαιωμάτων, να μας πούν τι συμβαίνει, ποια είναι αυτά τα έργα, τι προσπάθειες έχουν κάνει και να χρησιμοποιούν και τις εταιρείε συλλογική διαχείρισης. Είναι, πολύ, είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούν να έχουν το δικαίωμα αυτές οι εταιρείε να διενεργούν μια σοβαρή αναζήτηση σε ένα αρχείο, σε ένα μουσείο των κατόχων. Είναι αναγκαία να προστατεύσουμε επίσης τη διαδικασία web streaming, ε, χωρίς να την εμποδίζουμε. Ε, πολλές φορές μέσω του web streaming και της εμφάνισης ε, στο διαδίκτυο ε, παραβιάζονται δικαιώματα κατόχων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει και αυτό να το προσέξουμε. Ε, έχω τρεις εκπροσώπους της Κομισιόν. Ποιος θα μιλήσει παρακαλώ, η κυρία... Η κυρία, δεν ξέρω το όνομά σας. Πώς λέγεστε? Ποια είστε? Η κυρία Φερνάντες. Όχι. Είμαι η επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσωπώ την DG Markt, η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόταση αυτή και συνεργαζόμαστε βέβαια με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στο σχέδιο αυτοοδηγίας. Με την άδειά σας θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τα σχόλια που γίνανε. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ακριβώς ποια είναι η βάση της πρότασης αυτής. Δεν είναι μία πρόταση την οποία κάναμε επειδή έπρεπε να επινοήσουμε κάτι ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνων συζητήσεων που γίνανε με τους ε, φορείς που διαχειρίζονται ορφανά έργα, όπως οι βιβλιοθήκες, όπως ε, έργα διατήρησης και αποθήκευσης κινηματογραφικών έργων. Ήρθαμε σε επαφή με μεγάλα σημαντικά σχέδια όπως η Ευρωπαϊκή, οι διαδικτυακές βιβλιοθήκες και ζητήσαμε ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πρόταση προκειμένου να επιληθεί το γενικότερο ζήτημα των ορφανών έργων. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την πρόταση οδηγίας. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε γενικά και αόριστα για την συλλογική διαχείριση. Δεν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αποζημίωση των δημιουργών που δεν υφίστανται πλέον. Ουσιαστικά θέλουμε να απομπλεκάρουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά η οποία αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένη σε διάφορα ιδρύματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το όλο αυτό πλαίσιο και να καταλάβουμε και το μηχανισμό τον οποίο προτείνουμε. Είπαμε ότι θέλουμε να διευκολύνουμε την χρήση αυτή προκειμένου να καταφέρουμε να απελευθερώσουμε τα έργα αυτά Ξέρετε ότι πολλές φορές για διάφορα ντοκιμαντέρ του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου ή μπορώ να σας δώσω και άλλα παραδείγματα, θα μπορούσα να φερθώ και διάφορα βιβλία για τα οποία ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι. Πολλές φορές είναι έργα τα οποία γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι να πούμε το εξή Αν οι δικαιούχοι καταφέρουν καλή την πίστη να συνεργαστούν και αν καταλήξουν τελικά στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν τον κάτοχο των δικαιωμάτων, τότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να, να μπορούν να δώσουν μια ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα έργα. Όταν χρησιμοποιήθηκε η πρόταση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε κατά νου όλα αυτά τα αρχεία, όλες αυτές τις βιβλιοθήκες που βρίσκονται στα κράτη-μέλη. Και αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τους κατόχους δικαιωμάτων. Και ουσιαστικά είπαμε ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Εσείς είπατε ότι, κοστίζει πάρα πολύ η ενδελεχής αυτής έρευνα. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται. Αν πάρουμε τα βιβλία, τα κείμενα, τότε η έρευνα αυτή μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Στο παρελθόν χρειαζόντουσαν πέντε ώρες, τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα σε πέντε λεπτά. Αν μιλήσετε σε διάφορα ιδρύματα που προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν διάφορα πολιτιστικά έργα ή πολιτιστικό υλικό, ουσιαστικά θα σας πούνε ότι μπορούν αυτά τα ιδρύματα να κάνουν την εντελεχή αυτή λεπτομεριακή ανάλυση. Εφόσον λοιπόν αυτή γίνει και γίνει γρήγορα, τότε έχουμε και μία νομική εξασφάλιση για, το, για την ελεύθερη αυτή πρόσβαση για τα έργα αυτά. Πιστεύω ότι η ενδελεχή σε αυτή η ανάλυση θα δώσει ένα, μια νομική βεβαιότητα. Ουσιαστικά, μέσω τη οδηγία αυτή δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα μέσα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την αδειοδότηση. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά πράγματα εδώ πέρα. Από τη μια λέμε στα κράτη-μέλη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δρόμο που σας δίνει αυτή η οδηγία, το σχέδιο οδηγίας σε αυτή τη φάση, ή μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα διοδότησης τα οποία υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη έχουν λοιπόν την επιλογή. Τα συστήματα διοδότησης τα οποία υφίστανται είτε πρόκειται για τις σκανδιναβικές χώρες, στα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, είτε πρόκειται για συστήματα τα οποία υφίστανται σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία όλες αυτές οι λύσεις αδειοδότησης δεν έχουν να κάνουν με τα ορφανά έργα. Έχουν να κάνουν κυρίως για βιβλία, για παράδειγμα, τα οποία δεν εκδίδονται πλέον. Έχουν να κάνουν με άλλες κατηγορίες έργων. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να προβλέπει ένα σύστημα ενδελεχούς ανάλυσης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δίνει μία άδεια χρησιμοποίηση συγκεκριμένων έργων. Γι' αυτό το λόγο εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να δώσουμε και μία δεύτερη εναλλακτική λύση. Μπορεί κάποιο να κάνει την ε, λεπτομερή ανάλυση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει το ορφανό έργο ή στη διαφορετική περίπτωση, και ιδίω αν μιλάμε για μια βιβλιοθήκη εναρχείο το οποίο διαχειρίζεται χιλιάδες ορφανών έργων, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο άλλος δρόμος, αυτός δηλαδή της εταιρεία συλλογική διαχείρισης και στη συνέχεια να δοθεί μια άδεια. Τα συστήματα αδειοδότησης, οι λύσεις αδειοδότησης δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα τον δικαιούχο ως έργο και Σα τα λέω αυτά προκειμένου να σα εξηγήσω για ποιο λόγο προτείναμε μια διαφορετική λύση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για ποιο λόγο το σύστημα το οποίο προτείνουμε δεν βάλει σε καμία περίπτωση κατά του συστήματος το οποίο υπάρχει ήδη σε κάποιες καθναδικές χώρες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να κάνει τα πολιτιστικά ιδρύματα να πληρώσουν για έργα για τα οποία αγνοούνται ουσιαστικά οι κάτοχοι δικαιωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα δικαιολογείται με τίποτα. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια σαφή διαφορά ανάμεσα στα ορφανά έργα και τα έργα αυτά τα οποία έχουν περάσει στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά πράγματα, για δύο ξεχωριστέ κατηγορίε. Τα έργα τα οποία βρίσκονται στο δημόσιο τομέα μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν. Σα τα λέω όλα αυτά προκειμένου να αποσαφηνίσω κάπω την λογική τη πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ ισορροπημένη πρόταση που γίνεται ουσιαστικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθεται στα συστήματα διοδότηση τα οποία προβλέπονται ήδη στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι θα λέγαν το ίδιο. Ω Θεέ μου. Εσείς που καταλάβατε τα πάντα, πείτε μας λοιπόν. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στην εκπρόσωπο της Επιτροπής. Μίλησε για τα ορφανά έργα και μίλησε για προϊούσα έρευνα. Μπορεί να μας πει τι ακριβώς εννοεί, μέχρι πού προχωράμε χρονικά και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει ε, diligent research Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για διεξοδική αναζήτηση, τι νόημα έχει να ξέρουμε κατά πόσο ένα έργο είναι ορφανό. Για να το διαπιστώσουμε θα πρέπει να κάνουμε έρευνες για να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι είναι ένα ορφανό έργο. Και εάν ε, ορίσουμε τους έχοντες δικαιώματα, θα πρέπει να δούμε πώς θα τους φορούμε. ας πούμε. Ότι ένας κύριος Σμιθ έχει δημοσιεύσει ένα έργο, αλλά από τότε που δημοσιεύθηκε δεν έχουμε ξανακούσει για αυτόν. Δημοσιεύθηκε κατά τη δεκαετία του 60, ε, άρα ακόμα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και βλέπουμε ότι οι εκδόσεις ας πούμε πτώχευσαν 20 ε, ε, χρόνια πριν. Πώς μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να ξέρουμε κατά πόσο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε δικαιούχους. Πολλές φορές ε, μπορούμε να βρούμε τους δικαιούχους στο διαδίκτυο. Διαφορετικά προσπαθούμε να το δούμε με τα κράτη-μέλη και έχετε και το παράρτημα όπου βλέπουμε ποιες είναι οι ενδεχόμενες πηγές. λέμε ας πούμε οι εκδόσεις, αλλά ας πούμε πτώχευσαν οι εκδόσεις, ο εκδοτικός αυτός ε, ε οίκος. Θα έρθω λοιπόν σε επαφή με το Δημόσιο Φορέα Διαχείρισης. Ε, ίσως η λέξη, το όνομα Σμιθ δεν είναι και τόσο εφευρετικό, βρείτε μου ένα άλλο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει δικαιούχος μέσα στα πλαίσια μιας ορθολογικής σκέψης καθαρά. Κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις στην Κομισιόν για ορφανά έργα, πάντα μιλάμε για αυτά τα κριτήρια. Okay. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. θα να ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι, άλλα μέλη που θέλουν να παρέμβουν, άλλοι ομιλητέ ε, και η προθεσμία για, τις, ε, για τα ορφανά έργα είναι 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι όπως πάντα. Προθεσμία τροπολογιών. Και ε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τις παραδοσιακές διαδικασίες για τις τροπολογίες και πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου και όχι στο γόνατο σε ένα φύλλο χαρτί. Λοιπόν, η κυρία Σάκε, θέμα 7, μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά τηλεδιακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα μιας ε, περίπλοκης συζήτησης που κάναμε μαζί με την Επιτροπή uh, Empowering Ήτρε, για αυτό το θέμα της τηλεδιακυβέρνησης. Ε, θέλουμε να επιβάλλουμε ένα σχήμα με λιγότερη ε, γραφειοκρατία, λιγότερο δαπανηρό και που να προσφέρει μια καλύτερη χρήση προγραμμάτων λογισμικού πληροφορικής. αυτά προσπαθώ να παρουσιάσω στην, ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης, γι' αυτό προτείνω να συμπεριλάβουμε και πληροφορίες πνευματικών ε, πολιτιστικών οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά επίσης ε, την ανάγκη τονίζω για ψηφιακό γραμματισμό και για την ε, παροχή της κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να γίνει εύκολη πρόσβαση για να μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να έχουν συμμετοχή αλλά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη δημιουργία κατάλληλων φορέων, πλατφόρμας για την ε, καινοτομική χρήση αυτού του λογισμικού ανοιχτής πηγής και για τις ε, επιχειρήσεις και για το κοινό. Ε, ζητούμε λοιπόν όπως σας είπα πάλι τη συμπερίληψη πολιτιστικών φορέων για να τα βοηθήσουμε στην ψηφιοποίηση των ε, πληροφοριών και των, στοιχείων, των δεδομένων. Και επίσης ε, ζητούμε την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτής πηγής για να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, ε, ε, ε, εκπαιδευτών, καθηγητικού, ακαδημαϊκού προσωπικού κλπ. Επιγραμμικές πλατφόρμες δηλαδή. Deals with... Και θέλουμε να ενσωματωθεί ο ψηφιακός γραμματισμός στα σχολεία από μικρή ηλικία, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο λογισμικό αυτό, ε, το οποίο να μπορούν και να το επεξεργαστούν εύκολα. Okay. Äh, Εντάξει, ευχαριστώ. Μαρίκε. Ε, υπάρχει κανένας άλλος που θέλει να μιλήσει, Σαμπίνε. Ε, θέλω και εγώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η Μαρή Σάκε μόλις τώρα όσον αφορά την δυνατότητα της ελεύθερης χρήσης της τηλεδιακυβέρνησης. Πρέπει ε, νωρίς ε, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης να γνωρίσουν τα συστήματα αυτά ε, οι πολίτες μας ή δυνατόν από μικρής ηλικίας. Και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την μονάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάβασα τις συστάσεις και θεωρώ ότι είναι ευθυγραμμισμένες με αυτό που και εμείς θέλουμε να πετύχουμε μέσω του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, του νέου σχεδίου δράσης. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις προτάσεις που γίνονται στο κείμενο. Όσον αφορά τα σημεία αυτά τα κεντρώνονται περισσότερο στην εκπαίδευση, Δυστυχώ ε, δεν είμαι αρμόδιο για θέματα εκπαίδευση. δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω ένα συγκεκριμένο σχόλιο, Πάντω, γενικά μπορώ να πω ότι οι συστάσει που γίνονται ευθυγραμμίζονται με, τις, με τους στόχους και τι προτεραιότητες του δικού μα σχέδιου δράση. και όπω είπατε και εσεί όντω συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν περισσότερε ψηφιακέ δεξιότητε. και αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της ε, δικής μας ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. πολύ, κυρία Μπενεραπάτου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Μου προκαλεί ανησυχία το ψηφιακό χάσμα. Δηλαδή, Μιλάμε όλο και περισσότερο για τη χρησιμοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά ξεχνάμε κάπως και το τμήμα αυτό της κοινωνίας, το οποίο ενδεχομένω να μην έχει πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες και αναφέρομαι φέρουμε κυρίως στην τρίτη ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό οι τεχνολογίε αυτέ, οι ψηφιακέ αυτέ υπηρεσίε να μην είναι προσβάσιμε μόνο στου μαθητέ στο σχολείο, αλλά και στους εργαζόμενους, εργαζόμενους αυτούς που έχουν μια επισφαλή θέση εργασίας, θεωρώ ότι η ψηφιακή αυτή πρόσβαση είναι και ζήτημα δημοκρατίας τελικά. Υπάρχουν όλο και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες μας υποχρεώνουν να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο, να επισκεφθούμε ιστοσελίδες προκειμένου να καταφέρουμε να αποφεληθούμε από αυτές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην αποκλείσουμε από τις υπηρεσίε αυτές και διάφορα τμήματα του πληθυσμού και να φέρουμε κυρίως τους πιο ηλικιωμένους. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, λέει η Πρόεδρος. Τα προγράμματα που έχουμε για την ε, διαβίω εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες και πιστεύω ακριβώς όλες αυτές, ε, όλοι αυτοί οι ακαδημαϊκοί φορείς για την, της τρίτης ε, ηλικίας προσπαθούν να ε, διδάξουν και την ψηφιακή τεχνολογία σε μεγαλύτερους ανθρώπους, μεγαλύτερους σε ηλικία δηλαδή αλλά και τα παιδιά. Και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε όμως ε, ότι εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία, δεν έχουν computers. όμω ε, οι εργαζόμενοι μπορούν ε, να υποφεληθούν μέσω του κοινωνικού ταμείου με τα προγράμματα της διαβίου μόρφωσης, των προγραμμάτων κατάρτισης, ε, πολλά γίνονται ήδη για την ε, διδασκαλία ή για την χρήση, διευκόλυνση χρήσης και πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Η κυρία Μπερζέρ. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή τη συζήτηση γιατί μου φάνεται σημαντική. Δεν κατάλαβα τι εννοεί η κυρία Μπενεραμπάτου εγώ είμαι υπέρ της πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία διότι έχει μεγάλη σημασία να ακολουθήσουμε αυτό που είπε και η κυρία Σάκ. Σύμφωνα όμως με τις πληθυσμιακές κατηγορίες η προσπάθεια δεν είναι η ίδια και το αριθμητικό δεν είναι πανάκια. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ δεν θα έχουν πρόσβαση σε αριθμητικά δεδομένα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκτός συστήματος όσα χρηματικά μέσα και να διαθέτει η κυβέρνηση. Υπάρχουν μέρη, πληθυσμιακές μάλλον κατηγορίες που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία. Ιδιαίτερα στις, ε, στις διοικήσεις ή στους πιο ηλικιωμένους υπάρχει αυτή η, η απομάκρυνση. Γι' αυτό θα πρέπει βεβαίως να αξιοποιήσουμε το ψηφιακό αριθμητικό, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα άλλα μέσα, διότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν έχει πρόσβαση. Ναι, είπαμε να μην προσπαθήσουμε να, κάνουμε κάτι καλό και να καταλήξουμε σε κάτι αρνητικό. Ε, η ψηφιακή τεχνολογία ανήκει πλήχα στη ζωή μας. Ε, αλλά το ίδιο πρέπει βεβαίως να φροντίσουμε και τη γειτονιά μας, την κοινότητά μας, τους συμπολίτε μας. Δεν είναι ότι θα, τα πάντα στη ζωή μας θα τα αναλάβει η ψηφιακή τεχνολογία. Απλώς εδώ θέλουμε να είναι ανταγωνιστική η τηλεδιακυβέρνηση ε, σε μια ψηφιακή ενιαία ώρα. Εδώ πρόκειται για την ενίσχυση αυτής της ε, τηλεδιακυβέρνησης. Και η κυρία Σάκε είπε ότι θέλει να απομακρύνει λίγο την τηλεδιακυβέρνηση ε, από τους ε, ε, αρμόδιους φορείς και να μεταθέσει περισσότερο και ε, την ευκολία χρήσης και πρόσβασης στους καταναλωτές, στους χρήστες και στους πολίτες. Αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Δεν ήρθασταν καν. Δεν ήσασταν εδώ. Θέλετε να παρέμβετε σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν παρακολουθήσατε τη συζήτηση της Μαρίκη. Αν, ε, αν έπρεπε να είμαι καλή δασκάλα θα σας έλεγα όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι δασκάλα και σας δίνω το λόγο. E, σας ευχαριστώ πολύ. Ακολούθησα την συζήτηση μέσω του web streaming. Θα ήθελα, μάλλον για άλλη μια φορά σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Θα ήθελα να στηρίξω την εισηγήτρια, την κυρία Σάκη. Μας έδειξε ότι κατάφερε να προτιμάσει μια πολύ θετική έκθεση, ιδιαίτερα θετική για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στηρίζω το όλο σχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς πολίτες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο και να επιτρέπουμε σε όλους τους πολίτες να χρησιμοποιούν την κοινοτική εσωτερική αγορά και θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Σάκη, θέλετε να απαντήσετε να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο για τη συμβολή τους και θα ήθελα να καθησυχάσω όσους αναφέρθηκαν σε δημοκρατικό κίνδυνο. Η γνωμοδότηση αυτή θέλει ουσιαστικά να εκμεταλλευτεί τις δημοκρατικές ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία και η ψηφιοποίηση και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι χρειάζεται ψηφιακό γραμματισμός και εμπιστοσύνη προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένη και προσβάσιμη ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία θα καθιστά δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών. Τονίζω λοιπόν ότι η συμπερίληψη των πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του κειμένου. Η επί της ουσίας επιτροπή η ΙΤΡΕ θέλει να υιοθετήσει την έκθεση το Δεκέμβριο. Προθεσμία τροπολογιών 12 το μεσημέρι ε, στις 11 Οκτωβρίου. 11 Οκτωβρίου παρακαλώ, 12 το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν ως προς την ε, συνεδρίασή μας και τώρα και κλεισμένων των θυρών ε, η συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο πρωί στις 9 θα γίνει ψηφοφορία. Έχουμε ψηφοφορίες. Οι συντονιστές παρακαλώ να παραμείνουν. Βερονίκ, Ρομπέρτο.